πάνω από 20 συνεδρίες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αλφάνο. Λοιπόν, ευχόμαστε ε, καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Εχθές το βράδυ ο Προεδρεύων ε, στην Ολομέλεια ε, διάβασε μια ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 που πρότεινε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 4, καθώς δεν λάβαμε καμία αντίρρηση προσβολή αυτής της ε, ερμηνείας, εγκρίνεται η ερμηνεία. Τώρα ερχόμαστε στις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι. Ψηφίζουμε την έκθεση του κυρίου Μορέιρα. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κυργισίας. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία.